So, dear colleagues, welcome. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση αυτή. Καλώς ορίσατε, Πίτροπε Φεσχάγκερ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πριν να αρχίσουμε το διαρθωμένο διάλογο για τον ανταγωνισμό, έχω... Καταρχάς πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Σας ευχαριστώ και μετά έχω κάποιες ε, σύντομες ε, παρατηρήσεις για συνεχιζόμενους διαλόγους για το benchmark στις 23 με 25 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την πρόταση τροποποιητικού κανονισμού μια προσωρινή συμφωνία επετεύθη επί της ιδέας ε, των ε, benchmark για την μετάβαση ευρωπαϊκή μάλλον ε, κλιματολογική μετάβαση μετά πληροφορίες συγκεκριμένε θα περιλαμβάνονται στη δήλωση benchmark καθώς και αναχώρα benchmark. Οπότε συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την Νίνα Γκίλ. Τα καλυμμένα ομόλογα στις 26 συμφωνήσαμε για τους κανόνες περί καλυμμένων ε, στοιχείων και τους όρους για την οδηγία που θα πρέπει να τηρούνται ώστε τα ομόλογα να είναι επιλέξιμα για ειδική μεταχείριση τους ε, όρους για την ε, ε, δομή ολοκληρωσής τους και για την οδηγία που ήταν κομμάτι της Γενικής Διαπραγμάτευσης. Τεχνική εργασία έχει μείνει. Συγχαρητήρια στον κύριο Ρούκη και την διαπραγματευτική ομάδα. Επίσης, εργαζόμαστε πολύ σκληρά για την αναθεώρηση των επενδυτικών ε, εταιριών. Είχαμε διάφορους ε, τριμερείς στη διάρκεια της νύχτας. Ε, είχαμε τις τελικές διατάξεις. Οι τελευταίες συμφωνήθηκαν ώστε να εξασφαλιστεί ισότιμο πεδίο ανάμεσα στις μεγάλες συστημικές εταιρείες και τις μικρότερες επενδυτικές εταιρείες. Όλες θα διέπονται από το καθεστώς ε, προστασίας, οι κανόνες αντιστοιχίας για, για επενδυτικές εταιρείες τρίτων χωρών επίσης συμφωνήθηκαν πέρα από τις ε, διατάξεις θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες συστημικής σημασίας προς την Ένωση μόνο μετά από λεπτομερή αξιολόγηση από πλευράς της Κομισιόν με σημαντική και εποπτεία από την ΕΣΜΑ. Οι διαπραγματευτές επίσης ε, συμφώνησαν για τις διατάξεις διαφάνειας σε σχέση με τις επενδύσεις και τη συμπεριφορά του στη διάρκεια των συνεδριάσεων των ε, μετόχων. Ε, τέλος, θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρχουν συστηματικοί έλεγχοι στις 28 Φεβρουαρίου ε, συζητήσαμε και προοδεύσαμε Όσον αφορά την ε, αποκάλυψη βιωσιμότητας, επόμενος τριμερής θα γίνει αυτή την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Τέλος, ε, έκθεση SS 27 Φεβρουαρίου συζητήσαμε για, όσον αφορά τις διατάξεις για το ξέβλημα χρήματος. Η πρώτη ε, πολιτική συζήτηση για τις κοινέ διατάξεις για την ΕΖΑ για τη διοίκηση και τα λοιπά, αλλά δεν σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος ε, για την ΕΖΑ είπαμε ότι μια συμφωνία μόνο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος δεν θα είναι αποδεκτή, ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα ζητήματα. Αυτό σημαίνει πως το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο στην προσέγγιση του. Η Κομισιόν ζητήθηκε να συντάξει συμβιβαστικέ προτάσεις και η επόμενη συνεδρίαση έχει σχεδιαστεί για τις 12 Μαρτίου. Πολύ τριμερής λοιπόν, πολλή δουλειά, αλλά τώρα μπορώ να προχωρήσω τέλος στον δομημένο, διαρθρωμένο διάλογο με τη Μάργαρετ Φερστάγκερ. Πολύ μεγάλη χαρά μας που είστε σήμερα εδώ και όλοι γνωρίζουμε πως έχουμε συζήτηση για την πολιτική ανταγωνισμού. Είναι με προτεραιότητά μας και θέλω να εκφράσω την στήριξή μου στην εξαιρετική εργασία που έχει κάνει η Επίτροπος Βεσχάγερ. Δεν νομίζω πως υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στι βιώσιμες ισχυρές διατάξεις περί ανταγωνισμού και την προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού βιομηχανικού φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο κάνουν λάθος. Βεβαίως προβληματισμός και εργασία χρειάζεται για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πώς οι κανονισμοί μας θα εφαρμοστούν καλύτερα στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, αλλά αυτό δεν έχει σχέση, δεν έχει καμία σχέση με το ότι ούτω ή άλλω εμεί πρέπει να εξασφαλίζουμε το δίκαιο ανταγωνισμό εντό τη Ένωση ω προπόθεση για την ανάπτυξη ε, για καλύτερους όρους για τους καταναλωτές και για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς αλλά και προς χάρη της ανάπτυξής μας εν τέλει. Ε, Γιάννη Γιάννη και πρόσφατα επίτροπε έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά, έχετε ενισχύσει ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βεβαίως αυτό θα πρέπει και να το συζητήσουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε τη δική σας εισήγηση. Μάργαρετ, Μάργαρετ, έχεις το λόγο. Well, thank you very much. Ευχαριστώ και για τις ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις που ήταν πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι αυτός ε, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε ο διαρθρωμένος μας διάλογας. Ε, ήταν ουσιώδης, με λεπτομέρειες, αλλά με ξεκάθαρο στόχο, ξεκάθαρη οπτική για το ποιος είναι ο στόχος μας, δηλαδή η εξυπηρέτηση των πολιτών. Το λέω που βεβαίω με λυπεί και λίγο το γεγονό αυτό, γιατί είναι η τελευταία μου φορά εδώ στην ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ. Γιατί εδώ και πέντε χρόνια είχαμε πραγματικά άριστες συζητήσεις με την Επιτροπή σας. Συζητήσαμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο θα επιτρέπει την δημιουργία θέσεων απασχόληση με κοινωνικά δικαιώματα χωρί ταυτόχρονα να, χωρίς να γίνονται υποχωρήσει ε, στην ε, αγορά που πρέπει να εξυπηρετεί του πολίτε ω καταναλωτέ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συζητητέ που μας έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το ταξίδι, τον ε, κύριο Σμιτ, τον Βέρνερ Λάγκεν, τον Τίμπορ Σάνι, τον Ραμόν Τρεμόσα και βεβαίως τον Μισελ Ραϊμόν επίση. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδει ε, εισηγητές που προέρχεστε προφανώ από διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. Ε, από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, έχετε διαφορετικές οπτικές, ε, προτεραιότητες ε, σε ό,τι κάνετε. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι συνεργαστήκαμε πάντοτε σε πνεύμα συνένεσης, ότι η ίση όρια ανταγωνισμού, ο δίκαιος ανταγωνισμός, ο θεμητός ανταγωνισμός αποτελεί θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω η διέσμευση αυτή, η προσήλωση αυτή να διατηρηθεί εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και στη νέα τη σύνθεση μετά τι ευρωεκλογέ. Στο μεσοδιάστημα βεβαίω ε, η Κομισιόν ε, συνεχίζει το έργο της. Ε, μιλάμε για τη δουλειά. Δεν μπορούμε προφανώς να πούμε στους συνομιλητές μας και στους εταίρους μας στον κόσμο ότι σταματάμε τη δουλειά γιατί έχουμε εκλογές. Όλοι οι κανόνες θα επιβάλλονται και θα εφαρμόζονται κανονικά και το επόμενο διάστημα. Και θα συνεχιστούν βεβαίως και οι συζητήσεις ε, στο μέλλον ε, που ελπίζω και για εσάς ε, να αποτελέσουν και θέματα συζήτησης με τους εκλογείς, με τους ψηφοφόρους τα τελευταία, τους επόμενους μήνες. Υπάρχει λοιπόν το, η προτεραιότητα της, του ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή και πώς συνδέεται αυτό το θέμα με τα δεδομένα και την πρόσβαση σε αυτά. Και θεωρώ ότι για όλο ένα και περισσότερους πολίτες ε, το πράγμα γίνεται και σαφές, αλλά ε, γίνεται και μια ανησυχία. Πώς δηλαδή οι επιχειρήσεις ή ε, οι οργανισμοί στους οποίους εργαζόμαστε χειρίζονται τα δεδομένα μας, πώς συνδέεται αυτό με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται βλέπουμε πως οι συγχωνεύσεις ε, ε, εταιριών με δεσπόζουσα θέση, ε, με μικρότερες εταιρείες, επηρεάζει την καινοτομία και αναλύουμε όλα αυτά τα, αυτά τα δεδομένα, όλα αυτά τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα οι online πλατφόρμες, που προσφέρουν και δικές τους υπηρεσίες, μπορούν ίσως να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Φυσικά ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός και στον κόσμο offline και εδώ ε, μπορούμε να βασιστούμε σε στέρεα θεμέλια. Ε, βρισκόμαστε σε ένα σημείο σήμερα ε, με ένα μεγάλο εμπορικό πλεονέκτημα στα μεταποιημένα προϊόντα. 70% του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη απασχολείται, ιστορικά, ιστορικό υψηλό και η ποιότητα των θέσεων εργασία είναι καλύτερη από ό,τι στι περισσότερε άλλε περιοχέ του κόσμου. Δεν λέω ότι όλα είναι καλά, αλλά έχουμε διανύσει πάρα πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε. Φυσικά πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμη, ιδίω για του νέου, στην αγορά εργασία και ευρύτερα, αλλά και πάλι. Επίσης αντιμετωπίζουμε προκλήσεις ε, και στην παγκόσμια, στις παγκόσμιες Αντιμετωπίζουμε χώρες και εταιρείε που δεν είναι προσιλωμένες στον ε, δίκαιο ανταγωνισμό και καθώς ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο διασυνδεδεμένος, όλοι μας οι πολίτες, επιχειρήσεις, αρχές επιβολής του νόμου, ανησυχούμε ε, όλο ένα και περισσότερο για το πώς θα τα καταφέρουμε αν οι όροι ανταγωνισμού στο παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι ε, η θεμητή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και να υπερασπιστούμε τα δικά μας συμφέροντα με εμπορικές άμυνες όταν οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές μας ε, ε, ενισχύονται με επιδοτήσεις ή όταν προσπαθούν να κάνουν dumping στην ενιαία αγορά με τα προϊόντα τους επιμένοντας ότι αν οι άλλες χώρες θέλουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις δικές μας αγορές ε, τότε θα πρέπει να μας παρέχουν και εμάς πρόσβαση στις δικές τους αγορές. Γιατί όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες δεν υπάρχει αυτή η συμμετρία σήμερα. Επίσης, θέλουμε να προωθήσουμε και μια παγκόσμια ατζέντα κατά των επιβλαβών επιδοτήσεων και έχουμε εξοπλίσει την Ευρώπη με νέα εργαλεία για το σκοπό αυτό. Πλέον μπορούμε με σοβαρότητα να ελέγχουμε τις ε, ξένες επενδύσεις για να δούμε αν επηρεάζουν την ασφάλειά μας. Έχουμε αυτό το νέο ε, εργαλείο ελέγχου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτό ελέγχουμε ε, πώς μπορεί, ε, για παράδειγμα, να υπάρχει, να υπάρχει και κρατική παρέμβαση από εξωτερικούς φορείς σε στρατηγικούς ε, τομείς. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το μέγεθός μας για να καταπολεμήσουμε σε όλο τον κόσμο τον αθέμητο ανταγωνισμό. Φυσικά η ισχύ μας εξαρτάται από τις επιμέρους δυνάμεις που έχουμε και ε, οι επιμέρους δυνάμεις μας είναι οι ανοιχτές αγορές και η συνεργασία μας βέβαια Η ενιαία αγορά επιτρέπει στις εταιρείε μας, είτε είναι μεγάλες είτε είναι μικρές, να δείχνουν τι μπορούν να κάνουν, τις, ικανά, τις ικανότητές τους, να οξύνουν τις επιχειρηματικές τους και ε, ιδέες και στη συνέχεια να τα καταφέρουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις και οι κανόνες της Ευρώπης επιτρέπουν στον, ε, στις επιχειρήσεις μας μάλλον να αναπτυχθούν όχι μόνο οργανικά ε, μέσω της εσωτερικής ανάπτυξης αλλά και με, τις, ε, με την εξαγορά άλλων εταιριών. Ε, εγκρίναμε πάρα πολλέ συγχωνεύσει. Ακριβώ γιατί δεν έβλαπταν, θεωρήσαμε, τον ανταγωνισμό. Συγχωνεύσει που δημιούργησαν μεγάλου Ευρωπαίου παίκτε όπω την Opel και την Peugeot, την Imbev και την SAB Miller, Siemens και Gamesa. Τα τελευταία δέκα χρόνια εγκρίναμε πάνω από 3.000 τέτοιε συγχωνεύσει, απαγορεύσαμε μόλι 9. Και για κάθε εταιρεία που θέλει να εγκριθεί η συγχώνευσή της υπάρχουν συνήθως πολύ κλάδοι και καταναλωτές που επηρεάζονται. Ε, προφανώς ε, χρειάζεται κάθε εταιρεία στην Ευρώπη να έχει πρόσβαση και σε πρώτες ύλε και σε ε, υλικά για να μπορεί να παράγει τα προϊόντα της. Όταν λοιπόν έχουμε ανησυχίες, είναι κανόνας όχι η εξαίρεση, οι ίδιες εταιρείες να προσφέρουν ε, λύσεις. Για παράδειγμα με την πώληση περισσοϊκών στοιχείων ώστε η συγχώνευση να προχωρήσει χωρίς να στρεβλωθεί ο ανταγωνισμός. Αυτό το Φεβρουάριο δυστυχώς απαγορεύσαμε τη συγχώνευση Siemens και Alstom. Και όπως είπατε και εσείς στην έκθεσή σας, η περίπτωση αυτή ε, απαιτούσε πραγματικά πολύ λεπτομερή έλεγχο. Οι εταιρείε θα μπορούσαν να είχαν πάρει την ε, έγκρισή μας για συγχώνευση αν είχαν προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα για να διασκεδάσουν τις ανησυχίες μας που αφορούσαν τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν πρότειναν ξεκάθαρα αντισταθμιστικά μέτρα, είτε για τα συστήματα σηματοδότησης των σιδηροδρομικών αξώνων, είτε για τα, τους ε, σειρμούς υψηλής ε, ταχύτητας. Και αυτά αφορούσαν και επηρέαζαν την ποιότητα και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους στόχους της φιλικής προς το περιβάλλον μεταφοράς που θέλουμε να προωθήσουμε. Και δεν φτάσαμε μόνο εμεί σε αυτό το συμπέρασμα. Σε αυτό το συμπέρασμα έφτασαν και αρχέ ανταγωνισμού, παίκτε τη αγορά, ε, καταναλωτέ, ανταγωνιστέ, συνδικάτα, ενώσει ε, του κλάδου. Και τα σχόλια που λάβαμε από αυτούς ήταν αρνητικά τόσο για τα συστήματα, συστημα, συστήματα σηματοδότησης των αξώνων και για, τα, για τους ήρμους υψηλής ταχύτητας. Εμείς πάντοτε ε, σκεφτόμαστε πώς οι κανόνες ανταγωνισμού μπορούν να συνεχίσουν ε, να ενισχύουν τις επιχειρήσεις μας. Και το κάνουμε αυτό και με ε, το, το πλαίσιο για τα προϊόντα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, γιατί έτσι μπορούμε να παραμείνουμε αυτόνομοι σε σημαντικούς τομείς που θα εξασφαλίσουν την αυτονομία μας ε, στο μέλλον. Το Δεκέμβριο, λοιπόν, ε, εγκρίναμε ένα project στην μικροηλεκτρονική ε, με βάση τους κρατικούς κανόνες, ξέρετε, τα μικροηλεκτρονικά αφορούν τα μικροτσίπ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ε, αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς σε συσκευές οικιακέ. Γι' αυτό το project η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσουν δημόσια στήριξη προκειμένου να ξεκινήσει περισσότερη ιδιωτική επένδυση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Μεγάλες εταιρείε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει, ερευνητέ, νεοπαγεί εταιρείε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι αυτοί που θα συμμετάσχουν σε αυτό το project θα ε, μοιραστούν τις γνώσεις τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε οι φορολογούμενοι ε, που στην ουσία χρηματοδοτούν όλο αυτό το project να αποκομίσουν και τα ωφέλη. Αυτό δείχνει πώς η επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού και η οικονομική και η βιομηχανική ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίσουν. Στις ε, πέντε εκθέσεις που συντάξατε εσείς για την πολιτική ανταγωνισμού, εδώ το Κοινοβούλιο προσδιορίσε ποια είναι η κοινωνική ε, ελευθερία της ε, ε, οικονομία της αγοράς. Ανοιχτός χαρακτήρας, πυκλομορφία, δίκαιε ευκαιρίε για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές σε ολόκληρο τον κόσμο. Και για μένα αυτό είναι πραγματική έμπνευση ε, που πρέπει να καθοδηγήσει τη συζήτηση μας. Γιατί όταν συζητούμε την βιομηχανική πολιτική, και την βιομηχανική μας στρατηγική πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή δεν θα αφορά μόνο τους λίγους, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχω μαζί σας σήμερα. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βεστάγκερ και όπως πολύ σωστά είπατε είναι ο τελευταίος δομημένος διάλογος που έχουμε οπότε θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες της Επιτροπής μας ε, για την πάντα επικοδομητική προσέγγιση σας για έναν ανοιχτό και διαφανή διάλογο με το Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε πως ε, είναι ένας περίεργος κλάδος ο ανταγωνισμός όπου τα προνόμια της Κομισιόν δεν είναι τα ίδια με άλλους ε, κλάδους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να βρεθεί το σωστό μέτρο η ισορροπία μεταξύ της διαφύλαξης αυτής της ιδιαιτερότητας και της ανεξαρτησίας που επίσης σχετίζεται με τον ανοιχτό πολιτικό διάλογο. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη. Γι' αυτό ακριβώς και εκτιμούμε τις προσπάθειές σας. Και όπως μας υπενθυμίσατε υπάρχουν ε, διάφοροι κρίσιμοι τομείς. Ε, σήμερα συζητάμε τις ε, συγχωνεύσεις βιομηχανιών και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της ε, ψηφιακής ε, φορολόγησης. Όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά και χαίρομαι που έχετε την στήριξη του Κοινοβουλίου και της ε, Επιτροπής μας. Ξεκινάμε τώρα με τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Πρώτος ο κύριος Τόμ Φαντακεντελάρε του ΕΛΚ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, βάλτε τα ακουστικά σας για να με ακούσετε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα, αλλά και όλες τις υπόλοιπες μέρες, όχι μόνο σήμερα. Υπάρχει επίσης ε, πριν από δύο εβδομάδες η λεγόμενη υπόθεση για τις αποφάσεις υπερβολικών ε, πλέον αζώντων κερδών όπως λέγονται και η Κομισιόν λέει πως ε, αυτές ε, δεν θα πρέπει να ισχύουν για πολυεθνικές που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις και με την απόφαση αυτή της Κομισιόν δεν θα έπρεπε να πληρώνουν οι πολυεθνικές ε, φόρους για τα διεθνή, το διεθνές κομμάτι των κερδών τους. Ε, λοιπόν, είχαμε εδώ πέρα ένα σύστημα στα κράτη-μέλη όπου είχαμε μεμονωμένες ε, περιπτώσεις και κρίση κατά περίπτωση. Λοιπόν, ξεκίνησε το Βέλγιο άρα κατόπιν να προσπαθεί να ανακτήσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε Όμως τώρα οι δικαστές του δικαστηρίου λένε ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται για ένα ε, γενικό σύστημα αλλά για μια πρακτική στην οποία η εφορία τελικά ασκούσε την διακριτική της ευχέρεια. Οπότε δεν είναι πρόκειτο περί ενός συστήματος αλλά περί διακριτικής ευχέρειας. Ε, γι' αυτό ακυρώθηκε η απόφαση της ε, Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου είναι η πρώτη λογική ερώτηση, αν θα προσβάλλετε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερον, ε, αναμένουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να δουν τι θα γίνει με αυτήν την απόφαση. Ε, ποια θα μπορούσαν να είναι τα αποτελέσματα της απόφασης αυτού του δικαστηρίου κατά την απόψη σας και τέλος αν θα επηρεάσει την πολιτική σας. Για την τελευταία ερώτησή σας όχι, δεν, ε, ε, δεν έχουν έρθει σε επαφή άλλα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ακόμα εξετάζουμε το τι συνέχεια θα δοθεί. Κάποια πράγματα όμως τα οποία σημειώσαμε στην απόφαση είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα ε, το θεμελιώδες επιχείρημα ότι η Κομισιόν μπορούσε, δεν μπορούσε να τα δει αυτά ως ζήτημα κρατικών ενισχύσεων. Και εδώ πέρα απόψη είναι σαφή η Κομισιόν μπορεί να εξετάσει αυτές τις περιπτώσεις. Το δεύτερο, αυτό το οποίο αναλύουμε αυτή τη στιγμή, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε εμεί ως ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε βασικά α, ως κάποια κριτήρια εισόδου και μετά για κάθε εταιρεία η οποία πληρεί αυτά τα κριτήρια ε, υπάρχει ε, μια φορολογική απόφαση. Οπότε το δικαστήριο το είδε ως έναν συνδυασμό, δηλαδή ένα σύστημα ή ε, μεμονωμένες περιπτώσεις που μετά θα έλεγαν το τι θα έπρεπε να γίνει. Αν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια εταιρεία χρηματοδότησης εντός του ομιλού. Οπότε, ακόμα εξετάζουμε την προσέγγισή μας γιατί όπως είπα υπάρχει αυτός ο διτός χαρακτήρας ε, και συστήματος όπως θεωρούσαμε εμείς και μεμονωμένων αποφάσεων όπως το θεώρησε το δικαστήριο. Οπωσδήποτε όμως θα επανέλθουμε με πληροφορίες στο Κοινοβούλιο όταν ληφθεί μια απόφαση. Σας ευχαριστώ Νίνα Γκίλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω αυτά τα οποία είπατε προς την κυρία Βεστάγκερ. Με μεγάλη χαρά συνεργαστήκαμε και πραγματικά ήσασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Και όπως και εσείς, είμαι και εγώ σε μια από τις τελευταίες μου συνεδριάσεις, αλλά ελπίζω να συνεχίσετε να συνεισφέρετε. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο πράγματα όσον αφορά την σωστή ερμηνεία των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Μιλήσατε στην παρουσίασή σας για την επιδότηση των χωρών και θα πρέπει να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη και θα γνωρίζετε ότι πολλά κράτη-μέλη ενισχύουν για μία συγκεκριμένη χώρα, την Κίνα και λένε ότι το επίπεδο των επενδύσεων από κινέζικες εταιρείε και το πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι εταιρείε που είναι ακόμα κάτι το αδιαφανές δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και αναρωτιέμαι εάν η Κομισιόν θα εφάρμοζε τέτοιους ε, κανόνες με πιο ενεργητικό τρόπο και προς άλλες ε, εταιρείες που βασίζονται σε τρίτες χώρες εάν ισχύει κάτι τέτοιο και όπως είπατε είναι σημαντικό οι καταναλωτές βεβαίως να έχουν το καλύτερο δυνατό για αυτούς ε, και βεβαίως αν υπάρχουν κάποια μονοπόλια θα πρέπει Και βέβαια όσον αφορά την παραπληροφόρηση και σε σχέση με τον Brexit, οι κανόνε περί κρατικών ενισχύσεων είναι πραγματικά από αυτού που έχουν υποφέρει περισσότερο. Και συχνά αναφέρθηκε ω λόγο για τον Brexit. Παραδείγματο χάρη λένε ότι θα είχαμε προβλήματα εάν θέλαμε να επανεθνικοποιήσουμε τους σιδηροδρόμους. Και γνωρίζω πω σε πολλέ ε, χώρε ε, υπάρχουν κρατικοί σιδηρόδρομοι Χωρί να παραβιάζουν του. Ε, κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα μπορούσατε εσείς ως Επίτροπος Συνταγωνισμού να κάνετε μια δήλωση και να ξεκαθαρίσετε αυτούς τους κανόνες για να έχουμε κάτι συγκεκριμένο για εμάς που συνεχώς αντιμετωπίζουμε την παραπληροφόρηση. Σας ευχαριστώ. Για το θέμα των επιδοτήσεων έχουμε μια στρατηγική διμερή, μια πολυμερή και μια είναι ε, πολυμερής και μια εσωτερική. Στο διμερές τμήμα έχω διάλογο με τους ε, Κινέζους ομολογούς για τις επιβλαβείς αυτές τις επιδοτήσεις γιατί νομίζω ότι στην Κίνα έχουν 130.000 ε, κρατικές επιχειρήσεις και είναι και ζήτημα στρατηγικών επιλογών. Δηλαδή ε, δεν μην παίρνουν όλοι οι ενισχύσεις, αλλά μόνο οι στρατηγικές επιχειρήσεις. Και για εμάς το θέμα δεν είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει κρατικές ενισχύσεις, αλλά προσπαθούμε να μην βλάπτουν τον ανταγωνισμό, να είναι θεμητό ο ανταγωνισμός. Αλλά προφανώς δίνονται πολλά δημόσια κονδύλια. Μεγάλο κομμάτι από αυτό δεν θεωρούμε καν ότι είναι κρατικές ενισχύσεις. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό όταν μιλάμε για γέφυρες, ε, δρόμους και τα σχετικά ή πηγαίνει κανονισμό της γενικής εξαίρεσης. Οπότε υπάρχει αυτός ο απευθείας ε, διάλογος, αλλά και στα πολυμερή φόρα. Προσπαθούμε ακριβώς να το προωθήσουμε. αλφός μου, η κυρία Σεσίλια Μάνστον, ε, με τους ε, Ιάπωνες και Αμερικανούς ομολόγους της, πιέζει τον ΟΠΟΕ να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Νομίζω είναι σαφές ότι μεταρρύθμιση του ΠΟΕ ε, δεν θα γίνει σε έξι μήνες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να χρησιμοποιούμε σωστά τα εργαλεία που έχουμε στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να... να επιβάλλουμε τους κανόνες μας ε, εκτός επικρατείας μας, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά τα εργαλεία, τα εμπορικά, αν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνο όσον αφορά τους ίσους όρου ανταγωνισμού. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που μπορούν να γίνουν. Βεβαίω μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτού, ειδικά όταν συμφωνούμε να το κάνουμε από κοινού. Η δεύτερη ερώτηση για τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως λέτε, σε αρκετές χώρες έχουμε δημόσιες επιχειρήσεις. οι σιδηρόδρομοι, ενέργεια. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι είμαστε ουδέτεροι ως προς την ιδιοκτησία. Μπορεί να είναι κρατικές, ιδιωτικές. Εμείς θέλουμε μόνο αν κάποιοι είναι κρατικοί να μην τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Να είναι μια εταιρεία δηλαδή η οποία θα είναι αυτόνομη και θα παρέχει υπηρεσίες στην αγορά και ευχαρίστως ε, θα μπορούσαμε να σας δώσουμε και μία απάντηση γραπτός ε, αν υποβάλλετε μία γραπτή ερώτηση ε, θα γίνει το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ECR ο κύριος Λούκε και θα δώσω και την προεδρία στην Νίνα Γκίλ για 10 λεπτά. Είναι η τελευταία σας συνεδρίαση και είστε οι πρεσβύτεροι στην αίθουσα. Κύριε Λουκέ. Γεια σας ε, κύριε Επίτροπε. Θα μιλήσω γερμανικά. Σας έστειλα μια επιστολή στις 29 Ιανουαρίου για το Nortel για την υπόθεση αυτή. Δεν την έχετε απαντήσει ακόμη. Εδώ και πέντε εβδομάδες. Είναι ε, συνηθισμένη ε, αυτή η χρονική περίοδος ε, Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω πότε, περιμένω, πότε θα μπορούσα να περιμένω μια απάντηση ε, και ελπίζω να είναι και μια ουσιώδης απάντηση γιατί και επίση ούτε αυτό είναι δεδομένο δεν το απευθύνω ως κατηγορία προσωπικά σε εσά, αλλά συχνά συμβαίνει και αυτό οπότε γρήγορα απάντηση και σας παρακαλώ ουσιώδης για το Nortel B Βάσει δημοσιευμάτων στον τύπο ε, η εταιρεία αυτή έλαβε μία ε, έγκριση για αύξηση κεφαλαίου από εμπορικές τράπεζες αλλά και από τα κρατήδια της Σαξονίας Άνχαλτ και την κάτω Σαξονία. Μιλάμε για μια ε, αύξηση κεφαλαίου κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από εμπορικές τράπεζες ενώ τα κρατήδια θέλουν να δώσουν ε, περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα φορολογουμένων. Η Κομισιόν το 2012 στην διαδικασία που είχε ακολουθήσει αποφάσισε ότι η αύξηση κεφαλαίου από εμπορικές τράπεζες ε, ε, μπορούν να, ε, μπορούν να θεωρούνται ως κρατική ενίσχυση όταν οι εμπορικές αυτές τράπεζες ανήκουν στο κράτος. Δηλαδή μιλάμε συνολικά για κρατική ενίσχυση ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, όλα, όλα αυτά, αν πρέπει να συναπολογίσει κανείς ότι και το 2012 είχε δοθεί μια κρατική ενίσχυση πολλών δισεκατομμύριων ευρώ, με συνολική λοιπόν ε, επιδότηση αν, περίπου 15 δισεκατομμύριων ευρώ. Τότε η δικαιολόγηση, η αιτιολόγηση ήταν ότι αυτό γίνεται για να ξαναγίνει ανταγωνιστική η Nord LB. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Μήπως ε, συμφωνείτε λοιπόν με την δική μου αξιολόγηση ότι πρόκειται για μια στρέβλωση του ανταγωνισμού καθώς ε, επιδοτείται μια κρατική τράπεζα η οποία προφανώς δεν είναι βιώσιμη. Μήπως τελικά ε, αυτό αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού ακριβώς γιατί και άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους κρατική επιδότηση πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτούς τους στρεβλούς όρους ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ε, καταρχάς να σα ζητήσω συγγνώμη που δεν έχουμε απαντήσει στην επιστολή σα και σα διαβεβαιώ ότι ε, θα είναι ουσιώδη η απάντηση που θα σα δώσουμε. Ξέρετε, κάποιε φορέ όταν δεν είναι πολύ ουσιώδη οι απαντήσει μα, είναι ακριβώ γιατί δεν μπορούμε, δεν έχουμε ολοκληρώσει εμεί τι διαδικασίε, δεν έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία, προκειμένου να είναι η απάντησή μα ε, ουσιώδη. Βεβαίω, ε, σημειώνω το αίτημά σα. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί ακόμη, γιατί πρέπει πρώτα οι γερμανικέ εταιρείε να μα πούνε πώ θέλουν να προχωρήσουν όταν η εποπτική αρχή, ξέρετε, ε, λαμβάνει το αίτημα ότι χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια. Τότε η τράπεζα πρέπει απευθύνεται στην αγορά. Αν δεν τα καταφέρει να, κατα... να λάβει αυτά τα κεφάλαια από την αγορά, τότε πρέπει να δει τι θα κάνει. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με τι γερμανικέ αρχέ και όπως γνωρίζετε και από δημοσιεύματα υπάρχει και μια ιδιωτική προσφορά αλλά και μια προσφορά από τράπεζες που ανήκουν στο κράτος. Αυτό δεν μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε αμέσως ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση. Αυτό όμως που ξεκίνησε για μας είναι ότι κάναμε μια ε, πολύ λεπτομερή ανάλυση, γιατί ξέρετε ο πρώτος κανόνας για τις κρατικές ενισχύσεις είναι αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται ε, για το κράτη. Αν υπάρχει κάποια κρατική παρέμβαση εδώ ή εκεί, τότε πρέπει κανείς να πει ε, ότι εδώ πρόκειται για μια απόφαση του κράτους για χρήση κρατικών ενισχύσεων. Είπα και μόλις στην κυρία Τζιλ ότι δεν μπορεί κανείς να, να είναι Μπορεί, κανείς να, μπορεί μια επιχείρηση να είναι στην ιδιοκτησία του κράτους, αλλά δεν θα πρέπει να πληρώνουν οι φορολογούμενοι τα όσα κάνει. Εγώ, εξ όσων γνωρίζω, σε αυτή την περίπτωση ε, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, οπότε έχουμε το χρόνο να κάνουμε αυτό που πρέπει για να εξασφαλίσουμε την, την ίση μεταχείριση. Γιατί οι τράπεζες έχουν διαφορετική μορφή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δική μα ευθύνη είναι να θεωρήσουμε ότι οι τράπεζε είναι το ίδιο όταν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και αν υπάρχει κίνδυνο ε, παράνομων κρατικών ενισχύσεων, τότε θα πρέπει με, σε κάθε λεπτομέρεια, να, με κάθε λεπτομέρεια να αναλύσουμε την ε, εκάστοτε κατάσταση ανεξάρτητα από το ιδιωτικό καθεστώ τη ε, τράπεζα. Ευχαριστώ για του φιλελεύθερου. Ε, θα μιλήσω ο κύριο Τρεμόσα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε Βεστάγκερ, σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας για τη συζήτηση και θέλω να σας ευχαριστήσω και για την άριστη συνεργασία που είχαμε τα πέντε χρόνια. Ήταν πραγματικά ε, πολύ εύκολα τα πράγματα. Εγώ ήμουν εισηγητής πριν από τρία χρόνια. Η πρόσβαση πάντοτε και οι επαφές με, με το επιτελείο σας ήταν πάντοτε εξαιρετική. Ε, τις εκθέσεις τις συντάξαμε, ήταν εξαιρετικές σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες ε, του Κοινοβουλίου με απότερο στόχο πάντοτε να βρίσκουμε και τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τους πολίτες, καταναλωτές και τις επιχειρήσεις μας. Πριν από πέντε χρόνια σας είχα απευθύνει ένα ερώτημα για την υπόθεση Google και ε, τελειώνω αυτή τη φοιτεία με το ίδιο ακριβώς θέμα γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την υπόθεση αντιτράστ κατά της Google είδαμε ότι ε, ε, σας έχουν απασχολήσει και οι αναζητήσεις που προσφέρει η εταιρεία Google όχι μόνο τις κλασικές αλλά και για θέσεις εργασίας, ε, χάρτες κτλ. Επίσης είδαστε στον τύπο ότι ε, η Facebook θέλει να συγχωνεύσει το Messenger και το WhatsApp και το Instagram. Και τέλος, ε, υπάρχει μια υπόθεση κρατικών ενσύσεων που αφορά την Αλιτάλια. Μήπως έχετε νεότερες πληροφορίες να μας δώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον σας. Well, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όντως ε, και εγώ ε, μπορώ να πω ότι η συνεργασία ήταν ανοιχτή και απλή για θέματα τα οποία σας απασχολούν έντονα και με συνέπεια, ε, ε, όπως και εσείς ας πούμε ασχολείστε με το θέμα της Google, είναι σημαντικό να έχουμε ε, σταθερότητα στη ενδιαφέροντα και στα θέματα που μας απασχολούν. Πέντε χρόνια μετά είμαστε στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της τρίτης ε, υπόθεσης Google. Ε, έχουμε πολύ εντατικές διαδικασίες ε, εργασίας με την Google για την υπόθεση σύγκρισης Είχαμε μία απόφαση εκεί για, για πάυση ε, αλλά η απόφαση επίσης θέσπιζε μια αρχή ότι αυτή η περίπτωση θα σήμαινε και η συμμεταχείριση. Είναι μια υπόθεση δηλαδή ότι προσπαθούμε να πιέσουμε την νομοθεσία ανταγωνισμού για να αποδώσει. Γιατί μετά από αυτές τις τρεις ε, υποθέσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε τόσο γρήγορα κινούμενες αγορές η διαδικασία μπορεί να πάρει χρόνο ενώ η κατάχρηση να συνεχίζεται για πολύ χρόνο και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη πίεση για να μπορέσει να επανέλθει ο ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη αγορά. Θα το δείτε αυτό αν, παρακολουθήσετε τη συζήτηση για την, για την πολιτική ανταγωνισμό στον ψηφιακό στην ψηφιακή εποχή, θα διαπιστώσετε πως έχουμε επίσης μάθει από τις υποθέσεις ε, της Google. Γιατί δεν έχουν να κάνουν αυτές μόνο με τα πορίσματα, αλλά και για το πώς λειτουργεί η ψηφιακή αγορά για το μέλλον. Και αυτό πιστεύω θα το, θα το συζητήσουμε και αργότερα. Για το Facebook δεν είναι η ίδια η ολοκλήρωση που μας απασχολεί για να δούμε πώς χρησιμοποιεί τα στοιχεία η Facebook. Θα γνωρίζετε πως πολλές εθνικές αρχές στην Ευρώπη ε, αρχές ανταγωνισμού ενδιαφέρονται. Είναι σημαντικό γιατί και το Facebook είναι και διαφημαστική εταιρεία και εδώ η χρήση των στοιχείων είναι πολύ σημαντική και η χρήση των στοιχείων, η πρόσβαση στα στοιχεία, στα δεδομένα, θα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ψηφιακών αγορών. Για την Αλτάλια, μάλλον το παρακολουθείτε και εσείς στενά, Γίνεται προσπάθεια πώληση. Τώρα όσον αφορά τι κρατικές ενισχύσεις δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε πόρισμα, σε συμπέρασμα. Ευχαριστώ σε ευχαριστώ. Εκ των Πρασίνων έχουμε τον Μισελ. Σας ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για τα πέντε χρόνια συνεργασίες ε, και όλους τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές νομίζω για τα θέματα του ανταγωνισμού τους εκφράζω. Εντάξει, μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να είναι στην αγορά και το τι ε, πρέπει να είναι η ρύθμιση μεταξύ φιλελευθέρων και πρασίνων, αλλά εάν ε, για το εάν πρέπει να υπάρχει αγορά η οποία θα ρυθμίζεται σωστά, νομίζω υπήρχε μία συμφωνία. Τώρα, τα τελευταία, τις τελευταίες 10 μέρες, 10-15 ε, μέρες υπήρχαν κάποιες κρούσεις από τον Γάλλο και Γερμανό Υπουργό Οικονομικών για την απόφασή σας ε, για την Άλμστομ και λένε ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού. Ε, δεν είπαν ότι πρέπει να διαλυθεί και να καταργηθεί για να μπορούν έτσι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες να σταθούν διεθνώς απέναντι στον κινέζικο ανταγωνισμό. Εάν ε, το ερμηνεύσουμε αυτό, σημαίνει ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού το οποίο προστατεύει τους ε, καταναλωτές αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τόσο μεγάλες εταιρείες που να μπορέσουν να επιβληθούν σε άλλες αγορές ε, σε χώρες που δεν είναι τόσο πολύ υπέρ του δεν έχουν τέτοιο δίκαιο ανταγωνισμού και βασίζονται περισσότερο στον προστατευτισμό. Αυτό σημαίνει, αν το σκεφτούμε, ότι θα εξασθενήσει ο ανταγωνισμός στην εσωτερική μας αγορά για να μπορέσουμε να έχουμε εταιρείε ε, ανταγωνιστικές διεθνώ. Ε, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό σε ευρωπαϊκή πολιτική ε, ανταγωνισμού. Και όταν το λέει αυτό η γαλλική ή η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά. Θα ήθελα λοιπόν την πολιτική σας εκτίμηση. Ήδη υπήρξε μια συνέντευξη που δώσατε στους Financial Times και πολύ σωστά είπατε ότι οπωσδήποτε θα αποτελέσει θέμα προσεχώς ο ψηφιακός τομέας Facebook, Google και τα λοιπά για να προωθηθούν ίσως κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες που θα αντιμετωπίζουν διαφορετικά ίσως τα προσωπικά δεδομένα. Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει τα επόμενα πέντε χρόνια η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσουν ε, αυτές τις ε, κρούσεις των εθνικών κυβερνήσεων για την ε, μεταρρύθμιση του δικαίου του ανταγωνισμού. Λοιπόν, όπως είπα, ελπίζω ότι θα πιέσετε για να έχουμε αποτελεσματικά εργαλεία όταν θα γίνουν τα πάντα ψηφιακά. Αλλά αυτό ακόμα αντικατοπτρίζει τις, την θεμελιώδη επιλογή, όπως λέτε, εάν έχουμε αγορές και έχουμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, θέλουμε και ε, δίκαιο ανταγωνισμό. Όχι μόνο επειδή μας αφορά ως καταναλωτές, αλλά αφορά και τους πελάτες στην αλυσίδα ε, δημιουργίας αξία και η ευρωπαϊκή οικονομία χαρακτηρίζεται από μεγάλες και μικρές και μεσαίε επιχειρήσει, 20 εκατομμύρια επιχειρήσει νομίζω συνολικά. Μόνο 50.000 από αυτές εντωμεταξύ έχουν πάνω από 250 υπαλλήλου. οπότε υπάρχει ένα πλέγμα επιχειρήσεων ε, που επιτρέπει μια ευέλικτη και ανθεκτική και καινοτόμο οικονομία. Αλλά όλοι χρειάζονται βεβαίω ε, να μπορούν ε, να λαμβάνουν τις ε, πρώτες ύλες τους με λογικές τιμές και με καινοτομία για να μπορούν να κοινωνήσουν και οι ίδιες. Οπότε εγώ θα πίεζα για αποτελεσματικά εργαλεία και στην ψηφιακή εποχή και αυτό βασιζόμενη στην στρατηγική επιλογή του δικαίου ανταγωνισμού. Νομίζω ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Είναι εκπληκτική η ευρωπαϊκή βιομηχανία, παράγει πολλέ δουλειέ. Έχουμε και εμπορικό πλεόνασμα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίω ότι τα έχουμε κάνει όλα. Προφανώ ε, απομένουν πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά στην συζήτηση αυτή η αφετηρία είναι ότι τα πράγματα ψηφιοποιούνται. Τα δεδομένα θα είναι μια διάσταση της κάθε επιχείρησης. Ε, οι πλατφόρμες, η καινοτομία είναι μέρος της λογικής πλέον της παραγωγής ε, αξίας, ε, όχι η απαγόρευση της συγχώνευσης Siemens Alstom, η οποία συγχώνευση θα μπορούσε να έχει συμβεί εάν είχαν επιληθεί τα προβλήματα του ανταγωνισμού. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν μια χαρά. Υπάρχει ανταγωνισμό στα μετρό, στα τραμ, στα τρένα τα Intercity. Αυτό το οποίο απέμενε ήταν η σήμανση στις ε, μεγάλε γραμμές ε, και τα τρένα υψηλή ταχύτητα. Και μπορεί ακόμα να επιληθεί. Αν δείτε λοιπόν την παγκόσμια αγορά, και εδώ πέρα συμφωνούμε ότι η αγορά είναι παγκόσμια, τίποτα δεν εμποδίζει τις εταιρείε να κάνουν μια κοινοπραξία, αν θέλουν να υποβάλουν ε, μια κοινή προσφορά σε διαγωνισμό. Και τίποτα δεν εμποδίζει το να κάνουμε περισσότερα για να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προορισμού. Αλλά η αδυναμία μα δεν είναι η νόμη μα περί ανταγωνισμού. Αυτό είναι κομμάτι τη δύναμη μα. και νομίζω ότι έχουμε πολλέ συζητήσει ε, μπροστά μα. Αλλά όπω προσπάθησα να πω και στην αρχή, νομίζω ότι το να έχουμε μια ισχυρή βιομηχανική στρατηγική και να επιμένουμε σε δίκαιο ανταγωνισμό είναι πράγματα που μπορούν να συνδυαστούν και όχι πράγματα τα οποία θα πρέπει να θεωρούμε ως ζητήματα μεμονωμένα ή ότι το ένα αποκλείει το άλλο. Ελπίζω λοιπόν τα επόμενα πέντε χρόνια να δοθεί μια όθηση έτσι ώστε η ψηφιακή αγορά θα είναι μια αγορά όπου τα πράγματα θα αλλάξουν γιατί θα πρέπει να εξυπηρετεί τους πελάτες. Σας ευχαριστώ για την Γκουέ Μιγγέλ Βιέγκας να ε, Στην Πορτογαλία, καρπός δεκαετιών ε, δημόσιων επανεπενδύσεων, η σιδηρόδρομοι μας ε, καταραίων και οι πορτογαλικοί σιδηρόδρομοι έκαναν μια, ένα δημόσιο διαγωνισμό για να αγοράσουν ε, τροχαίο υλικό. Όμως ε, το φθηνότερο υλικό ήταν το κινέζικο, China Railways Rolling Stock Corporations. Αυτοί αποκλείστηκαν όμως. Αυτοί είχαν ήδη πουλήσει υλικό στην εταιρεία μετρό της Λισαβόνας. Έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις. Πώς να εξηγήσουμε αυτά τα διαφορετικά κριτήρια. Η ίδια εξοπλίζει το μετρό του Πόρτο, λέει το Ρομιλτής, αλλά αποκλείεται από το διαγωνισμό για τους πορτογαλικούς σιδηροδρόμους. Και γνωρίζουμε ότι είναι ανάγκη να υπερασπίσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Απλώ δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτό το κριτήριο δεν εφαρμόστηκε στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είχε βιομηχανία κατασκευή ε, σιδηροδρομικού υλικού. Όμω το όνομα αυτή του κριτηρίου ανταγωνιστικότητα αυτό εγκαταλείφθηκε τελείω και καταστράφηκε η βιομηχανία αυτή. Ε, και τίθεται λοιπόν αυτό το ερώτημα από πλευρά των Πορτογάλων. Είναι εφόσον έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει την βιομηχανία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες, όλων των χωρών ή αυτή η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς προστατεύει κάποιες εταιρείες κάποιων ε, κρατών μελών γιατί εδώ μιλάμε για 30 χρόνια και αυτό που συνέβη ε, στην Πορτογαλία προκαλεί όλες αυτές τις αμφιβολίες. Ευχαριστώ. Δυστυχώς, νομίζω πως υπάρχουν πολλά αίτια όταν υποφέρει η βιομηχανία. Ένα εξ αυτών προφανώς μπορεί να είναι ότι η βιομηχανία αντιμετωπίζει αθέμητο ανταγωνισμό διότι οι ανταγωνιστές δίνουν, παίρνουν κρατικές ενισχύσεις. Ένα αίτιο είναι αυτό. Ένα όμως από τα πράγματα που νομίζω πως μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι είναι να πούμε τι ακριβώς επιθυμούμε και ένα από τα πράγματα που η συνάδελφος Ρεσμπιέτα Καμκόφσκα ε, στηρίζει διαρκώς είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ σωστότερα τους κανόνες για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Γιατί εάν περιοριζόμαστε στο να βλέπουμε πόντους, εντάξει, τότε εκεί θα ανταποκριθούν οι εταιρείε. Αν όμω πούμε ταυτόχρονα ότι ναι, εντάξει, η τιμή είναι σημαντική, γιατί εφόσον πρόκειται για δημόσια επένδυση στο σιδηροδρόμου, στα τρένα, τελικά ο φορολογούμενο είναι αυτό που πληρώνει. Αλλά θα πρέπει να δούμε και την ποιότητα του προϊόντος, πόσο στο μέλλον θα μπορεί να ανανεωθεί, να εξυπηρετηθεί στο μέλλον, να διορθωθεί, να επισκευαστεί και η τιμή της επισκευής θα λαμβάνεται επίση υπόψη και όχι μόνο η αρχική τιμή της επένδυσης. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Εάν το κάνουμε αυτό τότε έχουμε πολύ πιο πλήρη εικόνα του συνόλου του κόστους της ε, δεδομένης επένδυσης και έχουμε και περισσότερα στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τον, οι οποίοι έχουν στόχο να δώσουν το φθηνότερη επένδυση αρχικά αλλά τελικά δεν συνεχίζουν να εξυπηρετούν αυτή την επένδυση αργότερα. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες για αυτό για τις αποφάσεις αυτές που λήφθηκαν στο παρελθόν, αλλά είμαι βέβαιη ότι στο μέλλον θα είμαστε πιο συνεπείς στο να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε, ώστε να εξασφαλίζουμε τον ανταγωνισμό, ναι βεβαίως, αλλά ε, να είναι και δίκαιος αυτός ο ανταγωνισμός. Και έτσι, στο στην παγκόσμια αγορά, ελπίζω πως τώρα το Συμβούλιο είναι το που πλοκάρει, αλλά θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το ε, διεθνές μέσο επενδύσεων, ώστε να είμαστε βέβαιοι πως όσοι έρχονται και συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς να ε, εξασφαλίζονται ότι υπάρχει αμοιβαιότητα, θα μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε στους δημόσιους διαγωνισμούς εκείνων των χωρών. Γιατί η ανοιχτή αγορά είναι πολύ καλή, αλλά είναι ακόμη καλύτερη αν είναι και συμμετρική. Και όχι μόνο μονόδρομη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάρκο Βάλη, Μάλιστα, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι, πριν από μένα θέλω να σας ευχαριστήσω Επίτροπε για την διαθεσιμότητα που δείξατε και την συνεργασία. Όμως να μείνω λίγο στην απάντηση που δώσατε στο συνάδελφο Λούκες για το κατά πόσο μια από τις επιλογές που υπήρχαν ήταν ότι η γερμανική αρχή δεν έχει δώσει ακόμα ε, τις επιλογές. Μία από τις επιλογές ωστόσο προβλέπει τη δημόσια συμβολή από πλευρά των Λάντερ ε, που εμπλέκονται. Βέβαια πρόκειται για δημόσια χρήματα και προφανώς αυτή η κατάσταση δεν ε, προβλέπει τίποτα το θετικό και για το περίφημο burden sharing που έχει αναφερθεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις, κυρίως στην Ιταλία όπου οι μέτοχοι χρειάστηκε να συμβάλλουν για την επίλυση της τραπεζικής κρίσης. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, δηλαδή αν χρειαστεί να εφαρμοστεί αυτή η προϋπόθεση από πλευράς του γερμανικού κράτους, η DG ανταγωνισμού θα ξεκινήσει επίσημη διαδικασία ή θα περιοθεί στο να, περιοριστεί στο να εγκρίνει αυτού του είδους την πρακτική και άρα να αμφισβητήσει αυτές που είναι οι ισχύουσες ε, διαδικασίες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ως γενικό μέτρο, διότι Είχαμε κάποιες αποφάσεις από το δικαστήριο που κατέστησε σαφές ότι η έναρξη διαδικασίας είναι η προτινόμενη η, προτιμόμενη μάλλον διαδικασία θα έχουμε μελετήσει και άλλες υποθέσεις και αυτό που είναι θετικό είναι ότι επιτρέπεται σε τρίτα μέρη να γνωστοποιήσουν τη θέση τους και σε επίσημη διαδικασία. Το άλλο είναι ότι θα είμαστε το ίδιο προσεκτικοί και εξονυχιστικοί σε αυτή την ανάλυση όπως και στις υπόλοιπες, διότι όπως λέτε όπως παρουσιάζεται τώρα και όλοι το γνωρίζουμε αυτό από δημόσιους ε, πηγές, Υπάρχουν δύο γραμμές πίστοσης, μία από τα δύο κρατήδια και ένα από την BACS. Και εδώ Είπα ότι θα είμαστε τόσο λεπτομερείς όσο και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί αυτό που αναζητούμε είναι βεβαίως είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να δούμε από πού κινούνται τα χρήματα για να δούμε αν αυτό θα μας δείξει κρατική ενίσχυση ή εάν τελικά είναι κάτι που κάποιος ιδιώτης επίσης θα μπορούσε να κάνει. Και αυτό είναι κάτι που εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε στην ανάλυση μας και βεβαίως θα είμαστε το ίδιο προσεκτικοί με τις γερμανικές τράπεζες όπως και με τις ιταλικές. Φυσικά η ίση μεταχείριση είναι θεμελιώδης αξία για το πώς λειτουργεί η Ένωση. Σας ευχαριστώ. you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για την ίση μεταχείριση που θεωρώ ότι θα απασχολήσει και την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το πλαίσιό μας, ιδίως όταν υπάρχει διαφορά και υπάρχουν διαφορετικά εθνικά καθεστώτα και υπάρχουν κενά στην νομοθεσία. Θα είναι μακρά ε, η συζήτηση Είχαμε άλλωστε και αντίστοιχη περίπτωση εδώ στο Κοινοβούλιο που συζητήσαμε επί μακρόν ε, θέματα ε, με το DGS ε, που κατέληξαν τελικά οι συζητήσεις αυτές γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο μπορεί να μην λειτουργεί πάντοτε στην εντέλεια αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο για τις μεγάλες τράπεζες για τις μικρότερες υπάρχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων που κατά τη γνώμη μου είναι και λίγο αντιφατικό. Ε, οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα, ένας τομής, ένας τομέας τον οποίο θα τον εξετάσει και θα τον συζητήσει η επόμενη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων με απότερο στόχο, όπως είπα, την βελτίωση του πλαισίου μας. Ελπίζω να καταφέρουμε να συνεχίσουμε το διάλογο με την Κομισιόν και για αυτά τα θέματα. Αυτά από μένα. Δεν βλέπω να υπάρχει ομιλητής από το ΙΕΝΕΦ, e οπότε ξαναδίνω το λόγο στο ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα της συνέντευξης που δώσατε στους Financial Times, όπου είπατε ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι που θα πρέπει να ε, κατοχυρώνεται από τα πάνω. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε παγκόσμιου ε, πρωταθλητές και να προωθήσουμε ευρύτερα την ε, εμπορική πολιτική. Μια και αναφερθήκατε λοιπόν στην εμπορική πολιτική, ποια είναι η γνώμη σας για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις εμπορικέ μα άμυνε, ιδίω όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων και πώ μπορεί να διαρθρωθούν αυτά. Ξέρετε ότι υπάρχει και σχετική συζήτηση που διεξάγεται και στο εσωτερικό των κρατών μελών γύρω από αυτά τα θέματα. Οπότε πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το δικό σα όραμα σε σχέση με την ε, πτυχή αυτή της πολιτικής. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια απέδειξαν ότι ο κόσμος ε, είναι όλο και πιο αλληλένδετος αλλά και πιο περίπλοκος. Η βιομηχανική πολιτική, η πολιτική ασφάλειας, η, εμπορική πολιτική διασυνδέονται όλο ένα και περισσότερο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ θα κάνω τα δικά μου και ας κάνουν οι άλλοι ό,τι ε, θεωρούν καλύτερο. Όχι, κάθε ένας ε, πρέπει να εντάξει τον εαυτό του σε μια ευρύτερη εικόνα. Γιατί όταν εμείς ορίζουμε κανόνες για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, για το πώς δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, τους λέμε να είστε έτοιμοι γιατί θα, θα δεχτείτε ανταγωνισμό. Γιατί αυτό είναι καλό για την καινοτομία, για τους καταναλωτέ κτλ. Όταν εμείς λοιπόν διατηρούμε αυτήν την πρόκληση στις ευρωπαϊκές αγορές, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε και στις παγκόσμιες αγορές. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Η συνάδελφός μου η Σεσίλια Μάλμστρομ προωθεί το θέμα αυτό πάρα πολύ, χρησιμοποιώντας τους αμυντικούς εμπορικούς μας μηχανισμούς. Τελευταία τέτοια περίπτωση ήταν και η αναθεώρηση αυτού του εργαλείου για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας. Γιατί και στο παγκόσμιο πλαίσιο, σε κάποιο, κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ε, ε, κάπως τυπολάτρες. Τώρα, πλέον, έχουμε πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες με ταυτόχρονη τήρηση πάντοτε των κανόνων. Και αυτό ε, ε, λειτουργεί και ως άμυνα και ως αποτροπή. Γιατί όταν τα πράγματα είναι, όταν εσύ ενεργείς πιο γρήγορα, ξέρετε, έχει, ε, ενισχύεται και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των κινήσεών σου. Όσον αφορά την ασφάλεια, όταν λέω ότι τα πάντα ψηφιοποιούνται, αυτό αφορά και την, το hacking, τις, την ασφάλεια, ε, την, ε, την κατασκοπία και εδώ ένα από τα στοιχεία για να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές είναι ε, η δυνατότητα που, που πρέπει να τους δοθεί να αξιοποιήσουν και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα ε, αξιοποιηθούν και στον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Το εργαλείο αυτό βεβαίως έχει μια περιπλοκότητα γιατί υπάρχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος αλλά υπάρχουν και εθνικοί κανόνες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ όλοι οι εμπλικόμενοι φορείς να εστιάσουν την προσοχή τους ε, σε αυτό το θέμα τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον για να τα καταφέρουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Νομίζω ότι είναι ανησυχία πολλών ανθρώπων. Όταν γίνονται επενδύσεις από έξω, αν οι επενδύσεις αυτές γίνονται για τα σωστά κίνητρα. Γίνεται μια επένδυση ακριβώς γιατί θέλει ένας επιχειρηματίας να δραστηριοποιηθεί σε αυτή την εξαιρετική ζώνη του, του πλανήτη, την Ευρώπη, ή μήπως για να πατήσει πόδι εδώ και να μας δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την ασφάλειά μας. Και είμαστε στην πολύ αρχή ακόμα, γιατί το εργαλείο αυτό ε, εγκρίθηκε και θεσπίστηκε πριν από λίγο καιρό. Γι' αυτό και οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι. Γιατί τότε, τους επόμενους μήνες δηλαδή, θα κληθούμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες που θεσπίσαμε. Και ξέρουμε ε, ότι το Κοινοβούλιο πλέον ε, οδεύει προς τη λήξη της θητείας του, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα εφαρμοστούν τα σημαντικά βήματα που έχουν αποφασιστεί. Ιδίω σε αυτού του πολύ ευαίσθητου τομεί, αλλά και σε άλλου τομεί. Όπου η εφαρμογή των κανόνων θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εξαρτή, αλλά και κατά τη διάρκεια τη συγκρότηση σε σώμα του νέου κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, εκείνοι που θέλουν να επανεκλεγούν, ε, επανεκλεγούν να πούν ότι εγώ ε, θα συνεχίσω να παρακολουθώ και ότι το έργο που κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματικά ε, τέθηκε σε εφαρμογή. Αυτό αφορά εμπόριο, ασφάλεια, ανταγωνισμό και ε, τις στρατηγικές μας αποφάσεις για το μέλλον. Γιατί διαφορετικά όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Σας ευχαριστώ. Μπαμπέτ Βίντερ. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω γερμανικά, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για όλα όσα μας είπατε. Είπατε ότι στο δίκαιο του ανταγωνισμού ο βασικός στόχος είναι η προστασία του πολίτη, του καταναλωτή και να εξασφαλιστεί ε, η ρύθμιση του ανταγωνισμού και στην ψηφιακή εποχή. Αυτά αφορούν και ερωτήσει μου. Αναθεώρηση του δικαίου των πνευματικών δικαιωμάτων που πλέον βρίσκεται στο στάδιο του τριμερούς διαλόγου και ε, θα έχουμε και την τελική ψηφοφορία μας εδώ στο Κοινοβούλιο το επόμενο διάστημα. Εγώ ε, ε, έχω παρακολουθήσει συζητήσει, έχω εργαστεί και στον τομέα του πολιτισμού και ξέρω πόσο δύσκολο είναι για τους, για τους εκδοτικούς οίκους, για τους συγγραφείς να διατηρήσουν τα έσοδά τους και την αμοιβή τους. οπότε για μένα το σύνθημα είναι ρύθμιση όχι απαγόρευση. Εγώ έχω λάβει χιλιάδες email για το θέμα των φίλτρων για το uploading ακόμη και αν δεν προβλέπεται έτσι ε, ακριβώς ε, στην ε, οδηγία αλλά εκφράστηκαν πολλές ανησυχίες για, το, για, το, για την οδηγία αυτή. Οι τεχνολογίες που κρύβονται πίσω από αυτές τις διαδικασίες ενέχει τον κίνδυνο να ενισχύσει έτσι περαιτέρω την ε, δεσπόζουσα θέση των μεγάλων εταιριών. Ακριβώς γιατί έχουν τα μέσα και τους πόρους για να αναπτύξουν τέτοια φίλτρα, ενώ οι μικρότερες εταιρείε δεν έχουν. Οπότε, από άποψη ε, ανταγωνισμού, οικονομικού, ε, ποια είναι η άποψή σας για αυτή την μεταρρύθμιση του συστήματος των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεύτερον, πριν από δύο εβδομάδες βρέθηκα στο πλαίσιο επίσκεψης της Επιτροπής ΕΚΟΝ στην Ιρλανδία και διαπιστώσαμε εκεί ότι η Ιρλανδία, το Δουβλίνο, έχει επωφεληθεί από τους ε, γίγαντες του διαδικτύου. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και ανησυχίες εν του Brexit ότι οι εξαγωγές της χώρας, της αυτής που συνήθως ε, με φυσικό τρόπο περνάνε μέσα από την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα τους δημιουργήσει εμπόδια ε, και ότι θα δημιουργηθούν ε, μεγάλα χάσματα μεταξύ υπαίθρου και πόλων στην Ιρλανδία. Και τρίτον, αν μου επιτρέπετε, ε, είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε από πολλούς ήδη. Εγώ βλέπω μια απόκληση αφενός ανάμεσα στην ποικιλομορφία στην Ευρώπη που είναι ευκταία, από την άλλη όμως και την ανάγκη να υπάρχουν αυτό που είπατε κι εσείς ε, ευρωπαϊκοί πρωταθλητές και δεν θα μιλήσω στους, ε, στους δρόμους αλλά για τα συστήματα με σηματοδότησης μια πραγματικά τεχνολογία εχμής η οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν μιλάω μόνο για την Γαλλία και την Γερμανία αλλά όπως και στην ε, Airbus θα μπορούσε αυτό το θέμα να αποτελέσει μια πανευρωπαϊκή επιδίωξη βιομηχανική. Um, Η μεταρρύθμιση του, δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, ξέρετε, δεν είναι στο χαρτοφυλακιό μου, αλλά με απασχολεί, γιατί δεν ξέρω κάποιον ο οποίος πάει στο YouTube για να δει τις ε, διαφημίσεις. Ίσως, ξέρω εγώ, για να δει τι γίνεται στο, τις διαφημίσεις στον τελικό του Super Bowl, αλλά με αυτήν την εξαίρεση πάνε για να δουν το, το κυρίως περιεχόμενο. Τα κλιπ τα διάφορα, τη μουσική, τις ταινίε, πράγματα που έχουν δημιουργήσει δημοσιογράφοι, ε, στιχουργοί, σκηνοθέτες, άνθρωποι με ταλέντο, αλλά βέβαιω αν δεν πληρωθούν πώς θα ζήσουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά επίγον να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Από την δουλειά την οποία εγώ βεβαίω παρακολουθώ εκ του Μακρόθεν ε, μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιόν νομίζω ότι ακριβώς το θέμα του μεγέθους και το ότι και εδώ έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις έχει συζητηθεί πολλές φορές Νομίζω ότι ο συμβιβασμός ε, τελικά είναι πολύ λογικός ε, στην περίπτωση αυτήν και είναι υπερβολή να πούμε ότι το παίρνουμε ε, ελαφρά και νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα επιτυχημένο συμβασμό. Δεύτερον, για το θέμα της Ιρλανδίας συνεργαζόμαστε με τις Ιρλανδικές αρχές για να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία που υπάρχει εντός ε, των κανόνων αυτών στο έπακρον. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύστημα που θα δίνει την εμπιστοσύνη ότι θα ελαφρυνθούν ε, οι επιπτώσεις ορισμένων καταστάσεων, ε, ειδικά αν υπάρξει ζήτημα που θα επηρεάσει τις ε, εξαγωγές. Γι' αυτό το έχουμε κάνει στην ομάδα εργασία, γιατί όπως ξέρετε η Ιρλανδική οικονομία είναι αυτή η οποία κινδυνεύει να πληγεί περισσότερο μετά το Ηνωμένο Βασιλείου και βεβαίως ε, είμαστε σε επαφή με τους Ιρλανδούς ακριβώς για να θα είναι ισχύει ότι έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία και υπάρχει και ένα σεμινάριο για τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται για να δούμε το τι γίνεται στο Ιρλανδικό πλαίσιο έτσι ώστε αν κράτη-μέλη βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση να δουν ε, ακριβώς ε, το τι έγινε στην περίπτωση της Ιρλανδίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ειδικά πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θεωρούν ότι υπήρχε κίνδυνος να βρεθούν ξεκρέμαστες. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό για τις ευρωπαϊκές ε, εταιρείε πρωταθλητές. Έχουμε αρκετούς από αυτούς και η συγχώνευση Siemens Alstom δεν ήταν μια συγχώνευση δύο ευρωπαϊκών μεγάλων εταιρείων, αλλά δύο παγκοσμίων μεγάλων εταιρείων όσον αφορά την τεχνολογία, το τι μπορούν να κάνουν στην σηματοδότηση των τρένων υψηλής ε, ταχύτητας ε, και παρά το ότι βεβαίως έχουν πολύ ικανούς ανταγωνιστές αν δούμε τους Ιάπωνες αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν υπάρχουν κινέζικα τρένα υψηλής ταχύτητας εκτός Κίνας εάν τα δείτε ε, θα είναι πάρα πολύ συχνά και Siemens ή Alstom τα κινέζικα τρένα ε, η διαφορά λοιπόν είναι ότι εδώ πέρα έχουμε ανταγωνισμό, ε, ενώ στην περίπτωση της Airbus είχαμε αρκετούς Αμερικανούς ανταγωνιστές, αλλά κανείς δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί στην Ευρώπη. Είχαμε μικρότερες εταιρείες που έφτιαχναν μικρότερα αεροπλάνα ή μέρη μεγαλύτερων αεροπλάνων. Και μετά όταν έγινε η συγχώνευση και προσπαθήσαμε να έχουμε την Airbus, μια ευρωπαϊκή εταιρεία, δημιουργήθηκε ο ανταγωνισμός. Οπότε οι δύο αυτές καταστάσεις είναι αρκετά διαφορετικές θα έλεγα, να μην πω αντίθετες. Είναι επίσης ε, σημαντικό να θυμόμαστε και να δίνουμε κατευθύνσεις για το πώς οι επιχειρήσεις όπως η Siemens και η Alstom μπορούν να κάνουν κάποιες κοινοπραξίες εκτός της Ευρώπης. Γιατί αυτό γίνεται εάν χρειάζεται να έχουν τέτοια κλίμακα, τέτοιο μέγεθος. Σας ευχαριστώ, Μπεντ Λουκέ. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα της κυρίας Βίντερ συγκεκριμένα το άρθρο 13. Είπατε ότι δεν είναι αρμοδιότητά σας το... τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά μετά είπατε ότι έχει κάποιες επιπτώσεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού η μεταρρύθμισή του. Μετά είπατε ότι το συζητήσατε επί μακρόν, καταλήξατε σε ένα συμβασμό που θεωρείτε ότι είναι ισορροπημένος. Ε, το τι θεωρείτε βεβαίως δεν μου αρκεί. Ε, το εξετάσατε, ασχολήθηκε η Γενική σας Διεύθυνση για το αν όντως από τις σκοπιές, ε, τις ε, νομικές ε, και του δικαίου του ανταγωνισμού αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν δεν είναι επιβλαβή και θα έχουν τη δυνατότητα οι μεγάλες εταιρείε να απτύξουν τέτοια φίλτρα για το ανέβασμα ή και οι μικρότερες αν θα έχουν αυτή την ικανότητα. Δεύτερο, επανέρχομαι στην ε, Nord Elbe την ε, τράπεζα. Είπατε ότι θα τα εξετάσετε και θα μιλήσετε με τις ε, γερμανικές αρχές και θα το δείτε σε λεπτομέρεια. Με ποια σειρά θα γίνει αυτό πριν πληρωθούν κρατικές ενισχύσεις είτε άμεσα από την κάτω αξονία και τους Αξανάνχαλτ είτε μέσω της Ένωσης των ταμιευτηρίων χρειάζεται η έγκρισή σας πριν εκταμιευθεί το πρώτο ευρώ ή θα δοθούν τα λεφτά και αν ε, το κρίνετε εσείς αναγκαίο θα επιστραφούν. Επίσης, ποια κριτήρια έχετε για αυτήν την λεπτομερή εξέτασή σας, ε, γιατί βεβαίως ε, σημαίνει ότι και η τράπεζα για να χρειάζεται αυτά τα κονδύλια ε, υφίσταται χρονική πίεση. Η εάν ε, καθυστερήσετε και πολύ θα μπορούσε να υπάρξει μια στρέβλωση στον ανταγωνισμού. Τέλος, δεν σχολιάστε για την αρχή ε, Μπέιλιν. Είπατε ότι ε, το τι είναι κρατικέ ενισχύσει εξαρτάται και από τη μορφή που θα έχουν, αλλά υπάρχει εντύπωση ότι σε τραπεζικέ ε, κρίσει, σε τελική ανάλυση, τα λεφτά προέρχονται από το κράτο και η αρχή του Μπέιλιν φαίνεται να παίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο. Ε, αυτό δεν είναι ικανοποιητικό και δεν είναι δυνατόν πάντα να εφευρίσκεται κάποιος μηχανισμός ως κράτος ώστε να χρηματοδοτούνται οι τράπεζες και οι αρχές ε, εποπτείας να λένε «Ε, ναι είναι κρατικά λεφτά, είναι το φορολογούμενο αλλά δεν τα θεωρούμε εμείς ε, κρατική ενίσχυση. λοιπόν έχουμε δημιουργήσει τις δυνατότητες να υπάρξει και bail με την BRRD. Γιατί δεν το εξετάζετε. Όπως σας είπα, η οδηγία αυτή για την πνευματική διοκτησία δεν είναι δική μα αρμοδιότητα και δεν είναι η δική μα γενική διεύθυνση που θα κάνει την ανάλυση. Δεν ξέρω τώρα το τι συνέβη με το συμβασμό αυτό, αλλά θα ήταν περίεργο να κάναμε εμεί κάποια τέτοια ανάλυση, γιατί γνωρίζετε πως οι γενικές διευθύνσεις έχουν οπωσδήποτε ελέγξει ε, ενδελεχώς τις διάφορες τέτοιες προτάσεις για να είναι ισορροπημένες. Όταν μιλάμε τώρα για την ε, εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στις τράπεζες, προσπαθούμε οι αρχές να γνωρίζουν το τι θα απαιτηθεί ε, από πλευράς χρόνου για να γίνει μια ανάλυση και επίσης θεωρώ ότι όλοι σε αυτόν τον κλάδο γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε απλά να υποθέσουμε ότι ε, είναι συμβατές. Μπορεί αργότερα να ανοίξουν κάποιες ε, περιπτώσεις και μετά γίνονται τα πράγματα πιο περίπλοκα. Εάν αναζητείτε μία λύση χωρίς ενισχύσεις, ε, που εντάξει μπορεί καμιά φορά να χρειαζόμαστε γιατί είναι μια κρατική ενίσχυση σε μια επιχείρηση και συγκεκριμένα σε τράπεζες, αυτό θα έχει σοβαρέ συνέπειε, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την αναδιάρθρωση. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι χρονικό πλαίσιο χρειαζόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και όπως είπα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάποια περίπτωση. Είμαστε σε επαφή με τις αρχές για να γνωρίζουν το τι θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό το οποίο κάνουμε πάντα είναι ότι σεβόμαστε την πρόθεση των κρατών μελών. Τι λύσεις ε, εξετάζουν. Μια φορά λέμε ότι ε, αυτό δεν είναι δυνατόν, ποια είναι μια άλλη εναλλακτική θέση σας, γιατί το νόημα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων είναι να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν, αλλά με έναν τρόπο που θα είναι ίδιος για όλους και εμείς να τηρήσουμε την εντολή μας. Δηλαδή όταν δίνονται κρατικές ενισχύσεις, να εξακολουθεί να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Και κοιτώντας την τραπεζική κρίση και όλα τα λεφτά των φορολογουμένων που μοιράζονται, είναι εκπληκτικά ποσά, πραγματικά. Ε, και στη Γερμανία και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες. Πριν λοιπόν την πειραρδή και την αλλαγή της ε, νομοθεσίας ε, δόθηκαν πολλές κρατικές ενισχύσεις και τότε καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να μειώσουμε θεωρώ την στρέβλωση του ανταγωνισμού και μου είπαν ότι τις πρώτες ημέρες ε, της οικονομικής κρίσης ε, ε, η προκατοχός μου κάποιες φορές έπρεπε να πει ότι όχι, δεν είναι δυνατόν να διαφημίζετε ότι έχετε εγγύηση του κράτους. Γιατί έχετε εγγύηση του κράτους για λάθος λόγο. Γιατί χρειαστήκατε κρατική ενίσχυση, οπότε μπορείτε να το διαφημίζετε κιόλα. Γιατί ο ανταγωνιστής σας άλλο στηρίζεται στις δυνάμεις του. Και προφανώς δεν μπορεί να διαφημίσει κάτι τέτοιο. Οπότε η δουλειά που έγινε ήταν πολύ λεπτομερής, ε, γιατί στην αρχή εμφανίστηκαν διάφορα ζητήματα. όπου δεν ε, υπήρχε ε, στο επίκεντρο ο δίκαιος ανταγωνισμός και τώρα είναι περίπλοκα τα Όταν χρησιμοποιείτε το VRD για την τελευταία σας ερώτηση, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για προληπτική ανακεφαλαιοποίηση υπό πολύ αυστηρούς όρους και αν υπάρχει εξαίρεση βεβαίως ε, είναι θεμητό για μια χώρα να ζητήσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εξαίρεση εάν βεβαίως ε, πληρούνται οι όροι. Και τέλος εάν ε, το Συμβούλιο αυτό της διάσωσης λέει ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά τότε είναι θέμα εθνικής, εθνικού πτωχευτικού δικαίου να φροντίσει τα ζητήματα αυτά στο εθνικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Όντως, ε, το bail είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και άρα ε, είναι θέμα γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά μάλλον επειδή έχει, είναι εξαιρετικά άκαμπτο, γιατί Διαφορετικά είναι πολύ βαριά επιλογή με 8% χωρίς μετάβαση. Αυτό δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Αυτό όμω έχει να κάνει με τον νομοθέτη. Εμείς στην επόμενη θητεία αναθεωρούμε αυτή την οδηγία και πρέπει ε, να διορθώσουμε με ανοιχτό μυαλό και να μην πούμε να το χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο επειδή ε, το έχουμε φτιάξει. καλή ερώτηση λοιπόν και θα πρέπει να απασχολήσει την επόμενη θητεία. Ja, eh, Σας eh, ευχαριστώ. Το 5G θα είναι νομίζω η ραχοκοκαλιά της νέας οικονομίας φαίνεται αυτό και στις επιχειρήσεις ε, και παντού. Βεβαίω, δεν έχουν όλοι, δεν θα πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση στα ιδιωτικά μας ε, δεδομένα. Το θέμα λοιπόν, η συζήτηση ε, όσον αφορά την Κίνα και το 5G είναι πάρα πολύ έντονη και θα πρέπει να υπάρξει μια χρήση με τρόπο ασφαλή. Και ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα μέτρα ασφαλείας ε, θα πρέπει να μπορούν να είναι συμβατά και με την ε, λειτουργία της αγοράς. Πώς θα φροντίσουμε λοιπόν οι μελλοντικές τεχνολογίες αφενός να είναι ασφαλείς και ταυτόχρονα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνουμε ε, και εμείς στον αγώνα αυτό του ψηφιακού ανταγωνισμού για να έχουμε την καλύτερη και την πιο ασφαλή τεχνολογία του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που μας απασχολούν όλους νομίζω αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως είπατε, όταν μπούμε σε, στα 5G είναι άλλη κατηγορία γιατί εκεί ε, έχουμε και φτάνουμε σε βιομηχανική κλίμακα στην ε, διαβίβαση δεδομένων. Ε, διαφορετικός βαθμός λοιπόν ολοκλήρωσης μπορεί αυτό να σημαίνει επιρροή στο, στο σύστημα υγείας, στο σύστημα ηλεκτροδότησης, την αυτόματη οδήγηση και ένα σωρό άλλα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ασφάλεια ε, software και ε, hardware. Πολύ λεπτό ζήτημα. Και βεβαίως τα μέλη τα οποία είναι πολύ προηγμένα στις συχνότητες θα πρέπει να πούν σε αυτούς που αγοράζουν τις συχνότητες ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν με το 5G. Για τις εταιρείε που θέλουν όμως να συμμετέχουν στις συχνότητες, να, αγοράσουν τις συχνότητες, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τι είδους κριτήρια θα ισχύσουν όταν ε, θα εξοπλίσουν το software ε, και τους εξοπλισμούς τους που θα πρέπει να αγοράσουν κάπου αλλού για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ε, το σύστημα που θα ισχύσει, ποια θα είναι τα κριτήρια. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση ακριβώς όπως υπάρχει και μια εθνική διάσταση, διότι ένα από τα πολλά υποσχόμενα του 5G είναι ότι μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας το γεγονός ότι σε συνοριακές περιοχές πολύ συχνά η συνδεσιμότητα πάει στο μίνιμουμ ή εν πάση περιπτώσει κάτι που δεν είναι πολύ σταθερό. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι αν έχουμε καλύτερη συνδεσιμότητα Αυτό θα πρέπει να ισχύσει όχι μόνο για ένα κράτος αλλά για όλα. Όλα θα πρέπει να είναι βέβαια ότι ε, ε, ισχύει και ότι υπάρχει ασφάλεια. Άρα λοιπόν Προσπαθούμε να βρούμε τι είδου ε, συμβουλέ ε, ή συστάσει θα μπορούσαμε να κάνουμε προ τα κράτη-μέλη, ώστε να γίνει ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για όλα αυτά. Γιατί, όπω λέτε και συμφωνώ μαζί σα, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εμπιστευτούμε την ασφάλεια αυτή τη υποδομή. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε νομίζω πω οι πολίτε θα πούνε εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, διατηρώ τις αμφιβολίες μου και αυτό μπορεί να είναι αρνητικό για όλα αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Να έχουμε δηλαδή ε, την ψηφιακό κόσμο που θέλουμε. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε τα θετικά θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε τα αρνητικά. Και εδώ η εθνική με την ευρωπαϊκή διάθεση θα πρέπει να συνεργαστούν. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα όλες αυτές τις απαντήσεις που θα θέλαμε να είχαμε εδώ και καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος, ο τελευταίος μεν, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και μπορούμε να κλείσουμε τώρα αυτό το σημείο παρακαλώ, ναι, έχετε το λόγο, ναι. Εγώ θα ήθελα μόνο να το πω αυτό, γιατί πραγματικά εκτίμησα τη συνεργασία μας. Έχουμε πετύχει πολλά, πιστεύω, όχι μόνο στη συζήτηση για συγκεκριμένα θέματα, αλλά ε, για μένα η όθηση που έχει δώσει το Κοινοβούλιο, η πίεση που έχει ασκήσει το Κοινοβούλιο λέγοντας ότι πρέπει να επιταχύνουμε, να τα καταφέρουμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες από ε, τον αθέμητο αντιγωνισμό και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν πως έχουμε καταφέρει κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο, δηλαδή να ενισχύσουμε τις αρχές μας, ε, τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, ώστε να κάνουν και εκείνες πολύ καλή δουλειά στις εθνικές αγορές, ε, πως θα μπορέσουν ε, δηλαδή να έχουν την απαραίτητη πρόσβαση σε μαρτυρίες και ούτω καθεξής, σε αποδεικτικά στοιχεία και ελπίζω πως όχι μόνο εσείς αλλά και οι συνάδελφοι σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο θα το χρησιμοποιήσουν αυτό στην εκστρατεία τους για να να δείξουν ότι κάνουμε κάτι το χρήσιμο που έχει νόημα ε, μέσω της συνεργασίας μας για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού ε, την έλεγχο των εθνικών ενισχύσεων ώστε να λειτουργεί καλύτερα και πιο εύρυθμα η, εθνική, εσωτερική αγορά και ως προς αυτό ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεργασία και εγώ με τη σειρά μου. Thank Suspension. Σταματάμε για λίγα λεπτά.

Συνάδελφοι, είστε έτοιμοι να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Uh, so, just a second. Eh? <coughs> Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία δοκιμαστικά. Ψηφίζουμε για να δούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά. της ψηφοφορίας. Τέλεια. So we start... Λοιπόν, ξεκινάμε με την ψηφοφορία για το αποτέλεσμα του τριμμένου λόγου για την διασυνορική διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων. Πρώτον για τον κανονισμό με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε 22 υπέρ, 0 κρατά 5 εποχέ. Ωραία. Περνάμε τώρα στην οδηγία για το ίδιο θέμα, επίσης με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. της ψηφοφορίας, 23 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Σε Συγχαρητήρια στον κύριο Κλίνσον, συγητή μας. Και περνάμε στην ψηφοφορία για τον της οικονομισμού για το MIFID. Πρώτη από κοινού ψηφοφορία για την παράγραφο 1 και 2. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ομαδική ψηφοφορία για τις αιτιολογικές ε, αναφορές υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και ομαδική ψηφοφορία για τις ε, τηλεολογικές σκέψεις υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και επί του συνολικού του κειμένου ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία 22 υπέρ, 0 κατά, 5 εποχέ, εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη συνεδρίασή μας είναι κοινή συνεδρίαση Έκον Ένβη τον, τη Δευτέρα στις 11 Μαρτίου στις 7.30. Θα επιβεβαιωθεί θα επιβεβαιωθεί, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη και την 5η 21 Μαρτίου συνεδρίαση ΕΚΟΝ στις 9 το πρωί. Λήξη συνεδρίαση, σας ευχαριστώ πολύ. I, see you. No, okay, good. Meeting is closed. Exactly. We have tomorrow now. That's something missing. We have tomorrow a joint Econ Libe meeting on recent. Έχουμε κοινή συνεδρίαση και με την ΛΥΜΠΕ ε, για τις τελευταίες εξελίξεις στις πράξεις κατεξοδότηση για το ξέπλυμα χρήματος που δεν ε, αρέσει ιδιαίτερα στο Συμβούλιο. Οπότε είπαμε να το συζητήσουμε αύριο. Αύριο λοιπόν. Τι ώρα? 7 το απόγευμα. Κοινή συνεδρίαση με την ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ. Τώρα λίγη συνεδρίαση.